Mes chers collègues, bonjour. Allez. Le projet d'ordre du jour peut être adopté s'il n'y a pas d'objection et je tiens à... Αν δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις, θα ήθελα να σας πω ότι το σημείο που αφορά την έκθεση τελίσκα και Σαλίνη θα τα αλλάξουμε. Θα δούμε πρώτα την έκθεση Σαλίνη και μετά την έκθεση Τέλιτσκα. Γιατί ο κύριος Τέλιτσκα έχει άλλες υποχρεώσεις για να μπορέσει να είναι παρόν κατά την παρουσίαση αυτής της έκθεσης. Κύριε Κράμερ, θέλετε το λόγο ήδη από την ημερήσια διάταξη, την έγκρισή της. Αύριο θα ψήσουμε για τα δικαιώματα των επιβατών Αναβάλαμε την ε, συνεδρίαση. βρήκαμε συμβαστικέ λύσει στην προηγούμενη συνεδρίαση, οι οποίε έγιναν αποδεκτέ. Φυσικά τι συζητήσαμε και πετύχαμε καλά αποτελέσματα. Θα σα ε, δώσουμε μια ανακοίνωση την Παρασκευή για μια εναλλακτική συμβαστική λύση, για την οποία δεν έχουμε συζητήσει ακόμα και ουσιαστικά πρόκειται για τροπολογίε αλλά ο χρόνος ε, δεν ήταν αρκετό αυτός. Θα είχαμε σωστές τροπολογίες ε, εφόσον δουλέψαμε μαζί με την ΙΜΚΟ και όταν ψάχνουμε τέτοιες ε, συμβαστικές λύσεις κάπου χάνουμε, κάπου κερδίζουμε. Ήταν πολύ καλός ο διάλογος και έτσι τα καταφέραμε. Όμως ήταν μόνο δύο άτομα εκ μέρους τεσσάρων πολιτικών ομάδων. Και αυτό είναι αντίθετο με τη διαδικασία, κάτι που δεν το έχουμε ζήσει τα τελευταία 14 χρόνια. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να αλλάξουμε την ψηφοφορία, να μην υπάρξει ψηφοφορία, να μην γίνει και να προχωρήσουμε πρώτα στην εναλλακτική συμβαστική λύση, να έχουμε νέες προτάσεις ε, για τροπολογίες και προφορικές ε, ε της γιατροπολογίας και να περιμένουμε μέχρι την Ολομέλεια. Αυτό που έγινε είναι απαράδεκτο για όλους τους συμμετέχοντες γιατί τρέξαμε να προλάβουμε και τελικά δεν ε, έπαιξε κανένα ρόλο όλο αυτό. Γιατί οι συντονιστέ τελικά αποφασίζουν τι θα κάνουμε. Ευχαριστώ. Monsieur Kramer, merci. Κύριε Κράμερ, σα ευχαριστώ για τα σχόλιά σα. Θα είμαι απόλυτα σαφή. Άκουσα το μήνυμά σα γι' αυτό αυτό το θέμα θα το βάλουμε στην ημερήσια διάταξη απόψε στους συντονιστές. Είναι απαράδεκτο να μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες την τελευταία στιγμή. Θα το συζητήσουμε απόψε για την αυριανή ψηφοφορία, για τα δικαιώματα των επιβατών και θα γίνει διαβούλευση απόψε. Σας ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο σας που ήταν ε, ιδιαίτερα προσήκον. Εγκρίνεται λοιπόν η ημερήσια διάταξη. Τώρα ως προς ανακοινώσεις της ε, Προέδρου δεν υπάρχουν ανακοινώσεις. Ναι, η Πρόεδρος είναι παρούσα, αλλά δεν, ε, δεν, ε, δεν έχει ανακοινώσεις. δεν πολυλογούμε εδώ. Αρχίζουμε λοιπόν με τη γνωμοδότηση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών μέσα στα πλαίσια του πολιετούς 21-27. Και δίνω το λόγο στον Ντομινίκ Ρικέ, τον εισηγητή μας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για τη βραχνάδα της φωνής μου, αλλά Έχω μια ασθένεια μεταδοτική, ελπίζω να μου περάσει. Έχω αρρωστήσει λιγάκι, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, είχαμε 44 τροπολογίες πάνω σε αυτήν την τροπολο... ε, έκθεση προς την ε, Επιτροπή Προϋπολογισμού για να θέσουμε τα ζητήματα που θεωρεί η Επιτροπή Μεταφορών σημαντικά. Έγινε μια συνάντηση για να τα συζητήσουμε αυτά με τον ε, η εισηγητή, μία ήταν αρκετή, καταλήξαμε σε οκτώ συμβιβαστικέ. Οι οποίε καλύπτουν το σύνολο των θεμάτων της έκθεσης. Ε, όλες οι τροπολογίες την χάνουν της υποστήριξης ε, των πολιτικών ομάδων όλων, εκτός από την τροπολογία 3, στην οποία αντιτίθεται το ECR. Όλες τις υπόλοιπε λοιπόν τις τροπολογίες τις υποστηρίζουν όλοι, εκτός βέβαια από το ΕΝΕΦ e που δεν γνωρίζουμε ποια είναι η θέση του γιατί δεν εκπροσωπήθηκε στην συνάντηση των ε, σκιωδών. Φαντάζομαι ότι η έκθεση αυτή δεν θα δημιουργήσει προβλήματα διχογνωμίας γιατί αντικατοπτρίζει ανησυχίες όλων μας. Αυτό που είναι πιο δύσκολο είναι αυτή η μεταφορά κοντιλίων από το Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης προς το νέο μηχανισμό ε, ε, των ταμείων για τις μεταφορές. Αυτό είναι το μόνο. Σας ευχαριστώ κύριε Ρικέ. Πριν να δώσω του λόγο στους σκιώδεις, δεν θέλω να καλωσορίσω τους φοιτητές δημοσιογραφίας που μας επισκέπτονται και βρίσκονται στη Καλαρία, στην στο βάθος. Καλώς ορίσατε. Vous venez de quel pays? Από ποια χώρα προέρχεστε? De, de, vous venez d'Allemagne et des États-Unis? Γερμανία και Ηνωμένε Πολιτείε. Μάλιστα. Από παντού, από, από διάφορα μέρη του κόσμου λοιπόν. Εξαιρετικό. Βλέπετε που η Ευρώπη ανοίγει τις πόρτες της ολόκληρο τον κόσμο. Λέει η Πρόεδρος, καλώ ορίσατε και πάλι. Κύριε Βαντερκάμπ, έχετε το λόγο ως σκιώδης. Ε, ε, Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Ρικέ, Είχαμε εξαιρετική συνεργασία. Όμως, έχει υπάρξει ένα πρόβλημα, ένα λάθος που διαπιστώνω, κάτι που δεν καταγράφηκε σωστά στην ε, συνάντηση των σκιωδών. Είχα προτείνει ε, σε σχέση με την τροπολογία 3, σε σχέση με τη συμβιβαστική τροπολογία 3, να προσθεθεί μια διατύπωση να διαγραφεί μάλλον η διατύπωση accessible to all member states, να είναι προσβάσιμο σε όλα τα κράτη-μέλη. Είχα πει ότι αυτό δεν χρειάζεται, γιατί τα Ταμεία περιφερειακή ανάπτυξη είναι προσβάσιμα σε όλα τα κράτη-μέλη. Ο συνάδελφο που είχε υποβάλει αυτή την τροπολογία λέγοντας ότι βοηθάει στη σαφήνεια του κειμένου, αλλά εγώ είχα ζητήσει την Τετάρτη στη συνάντηση των σκιωδών να διαγραφτεί αυτή η φράση, μια και είναι περίτη. Κατά λάθο διαπιστώνω ότι αυτό δεν έγινε. Θα ήθελα να ζητήσω από τον Ντομινίκ και από το προσωπικό της γραμματείας να διορθωθεί αυτό. Η κυρία Ιζαμπέλα Ντεμόντε. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική εργασία, τον κύριο Ρικέ, καθώς και τις ε, προτάσεις συμβιβασμού που πάνε πολύ καλά. Έγινε μία συνάντηση, αλλά βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία του τουρισμού, γιατί όσο προχωράμε σε αυτή την εργασία, φτάσαμε σε μία σαφή αναγνώριση των θεμάτων και ευχαριστώ τον εισηγητή για τις προτάσεις συμβιβασμού. Νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια εγγραφή στον προϋπολογισμό για να μην υπάρχει κατακαιρματισμός των ε, κονδυλίων. Στη δεκαετή κρίση που ε, ζήσαμε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε η τρίτη οικονομία της Ευρώπης και αντισταθήκαμε αρκετά στην κρίση. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε μία αποφασιστική απάντηση αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες του τομέα του τουρισμού. Επίσης υποστηρίζω τον οργανισμό εργασίας που θα πρέπει να έχει τον κατάλληλο προϋπολογισμό για να μπορέσει να ασκήσει τα καθήκοντά της. Ευχαριστώ τους σκιώδεις, τους βοηθούς και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε μια θετική πρόταση. Ο κύριος Ζωτόσκι θα λάβει το λόγο εξ του κυρίου Ζήλε. Όχι, όχι, ωραία. Ο κύριος Κράμερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ την συγγύτρια. Έχουμε υποβάλει προτάσεις για υποτροπολογίες οι οποίες έχουν ενταχθεί όμως ε, στη συμβαστική πρόταση. Θέλω να ευχαριστήσω, δεν έχω να ασκήσω κριτική σε κάτι άλλο, οπότε ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Η κυρία Κιλόνεν από την ΚΟΕ, όχι. Ε, ο επόμενος ομιλητής, η επόμενη ομιλήτρια μάλλον η κυρία Νταλόν. Ευχαριστώ πολύ τον Ντομινίκ Ρικέ που παρόλο που είναι άρρωστος ε, σήμερα, είναι αρκετά μαχητικός έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις του στα πλαίσια του πολιετούς που είναι η μάχη των μαχών για να μπορέσουμε να ορίσουμε τα τομεακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί έχουν ε, υποβάλει τροπολογίες για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνδεσιμότητας ή για τον οργανισμό για τις δορυφορικές συνδέσεις με στα πλαίσια του πολιετούς. Και γι' αυτό υποστηρίζω την πολιτική θέση του εισηγητή έτσι ώστε να έχουμε 12,3 δις στα πλαίσια της ε, συνδεσιμότητας. Θα επαγρυπνούμε έτσι ώστε οι μεταφορές να μην είναι ένα τομέα ίσονος σημασίας. Επίσης, προβλέπουμε 20 δις στα πλαίσια των περιφερειακών διασυνδέσεων και θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί 10% του συνολικού ποσού για το ΕΤΠΑ. Εν πάση περιπτώσει θα θέλαμε να ενισχύσουμε τις μεταφορές στον περιφερειακό τομέα και να υπάρχει μια θεματική συγκέντρωση έτσι ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις επιμέρους συνδέσεις. Η κυρία Γκραπίνη. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, σίγουρα και εγώ θα συγχαρώ τον εισηγητή. Νομίζω ότι από τόσα συγχαρητήρια θα γίνει καλά θα ήθελα να πω τα εξής. Προβάλαμε τροπολογίες, έχουν υποβληθεί τροπολογίες οι οποίες δεν αρκούν για μια καλή συνδεσιμότητα. Μιλάμε για 12 και 13% μείωση του τομέα των μεταφορών και του Ταμείου Συνοχής. Αυτά δεν είναι θετικά. Γι' αυτό θα ήθελα να πω αυτά που είπε και η Ιζαμπέλ, δηλαδή εγώ τόνισα το τομέα του τουρισμού, ο οποίος ε, έχει αμεληθεί. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο Έχω υποβάλει και εγώ τροπολογίες, ελπίζω να ληφθούν υπόψη. Αλλά θα ήθελα να πω ότι αυτές οι μειώσεις για το νέο πι δελτα πι, θα, αυτές οι μειώσεις θα γίνουν αισθητέ γιατί ο κύριος Βαντεκάμπ ήθελε να αποκλείσει έναν ορισμένο τομέα και συγκεκριμένες περιφέρειες. Άλλαξε όμως γνώμη στη συνέχεια. Γι' αυτό θα πρέπει να μην πλήξουμε τους πολίτες. Υποστηρίζω την έκθεση, αλλά θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη για τα ε, ποσά αυτά και για να μην γίνουν περαιτέρω μειώσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ όλους τους ε, συναδέλφους, τους κοιόδης που έλαβαν το λόγο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ρικέ, τον εισηγητή μας. Γιατί αν με κολλήσετε κύριε Ρικέ και δεν έρθω αύριο, εσείς θα φταίτε. Το λέω. Έχετε το λόγο. Bien, euh, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους σκιώδεις για την καλή συνεργασία που είχαμε και τους συναδέλφους που πήραν το λόγο εδώ. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούσαμε στις ανησυχίες. Δεν είναι και κάτι δύσκολο. Δεν ήταν και τόσο δύσκολο να συμφωνήσουμε, γιατί σημείωσα ωστόσο την παρατήρηση του Βιμ. Εγώ θα πρότεινα. Αφού συζητήσατε να διαγραφεί αυτή η φράση, θα πρότεινα αν και δεν είναι και τόσο δόκιμο, αν θέλετε, ως διαδικασία, μιας και διαπιστώνω ότι όλοι συμφωνούμε, να γίνει η διόρθωση που ζήτησε ο ΒΙΜ με την άδεια κιόλας και της ε, Προέδρου και του Προεδρίου μας, να κρατήσουμε αυτή τη, ε, αυτή τη φράση όπως το είπε ο ΒΙΜ. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο απλό, γιατί όλοι συμφωνούν και βλέπω ότι γνέφεται όλοι με χαρά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εμεί ευχαριστούμε κύριε Ρικέ. Να υπενθυμίσω ότι η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στην Επιτροπή μας στις 9 η ώρα το πρωί. Και μπορούμε να συνεχίσουμε. Θα περάσουμε στο σημείο 5, δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής για την Εργασία είναι ε, γνωμοδότης ιδίας πρωτοβουλίας της ε, Επιτροπής Απασχόλησης και η κυρία Τέτιεν είναι, η... είναι ο μας. Ευχαριστώ. Η ασφάλεια της μεταφοράς είναι ένας καθοριστικός ε, τομέας για τη συνεργασία και την κοινή ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κανέναν άλλο κλάδο της οικονομίας είναι τόσο εξαρτημένη ε, η σωστή λειτουργία της Ευρώπης. Οι κανόνες για την ασφάλεια, ε, διασωρική συνεργασία και η κοινή, νομοθεσία για την εργασία ε, όπως ξέρετε, για τον έλεγχο των βαρέων οχημάτων. Ως ε, βουλευτές πρέπει να έχουμε στόχο η νομοθεσία να εφαρμοστεί στον χώρο της εργασίας. Σε πολλές μελέτες καταλήγει η Επιτροπή ότι οι ισχύουσες διατάξεις στον τομέα της μεταφοράς είναι διαφορετικές, εφαρμόζονται διαφορετικά. Όσον αφορά τον έλεγχο, τον, τους οδικούς ελέγχους, ε, υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις σε αυτές τις διατάξεις. Υπάρχουν ε, Διαφορέ πάρα πολλέ για έναν τομέα που είναι από του πιο σημαντικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι δύσκολο και για τι επιχειρήσεις και για του εργαζόμενου. Ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εργασία θα προσπαθήσει να εναρμονίσει τι συνθήκε εργασία σε όλη την ε, Ευρώπη και εν ονόματι του ε, ισότιμου ανταγωνισμού θα προσπαθήσουμε ε, μέσω αυτού του οργανισμού να βελτιώσουμε την νομοθεσία. Στην γνωμοδότησή μου για τον, οργανισμό αυτό τονίζω ότι ο ε, οργανισμός αυτός θα ε, συμπληρώσει ένα κενό, ότι δεν είναι μία ε, δομή η οποία θα επικαλύψει στις δραστηριότητε κάποια άλλη. Θα πρέπει να υπάρξουν ε, καλύτερη και πιο αποτελεσματική έλεγχη και σωστή συνεργασία μεταξύ των ε, εθνικών αρχών, ώστε να υπάρχει και καλύτερη ιδιαιτησία και διαμεσολάβηση σε περίπτωση διαφορών. Τα συστήματα που υπάρχουν μέχρι στιγμής θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και να επεκταθούν προς όφελος των εργαζομένων. Το European Road Register για τις μεταφορές, όπου ε, υπάρχει η πρόσβαση σε διασύνδεση εθνικών ηλεκτρονικών μητρών επιχειρήσεων μεταφορών. Επίσης, η οδική έλεγχη που θα πρέπει να λαμβάνουν χώρο ώστε να μπορέσει ο οργανισμός αυτός να βοηθήσει τις εθνικές αρχές. Επίσης την εκπαίδευση των ελεγκτών της οδικής κυκλοφορίας. Χαίρομαι ότι έχουμε υποστήριξη και στα άλλα κόμματα για αυτά τα σημεία που προτείνουμε. Σήμερα η Επιτροπή Μεταφορών ε, μπορεί να στείλει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα ώστε να υπάρξει ισότιμο συνταγωνισμό στον τομέα των μεταφορών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Σιγητά, Ευχαριστώ για την πολύ καλή συνεργασία, για το ότι είστε ανοιχτό σε προτάσεις. Θα ξεκινήσω λέγοντα ότι κάνουμε λόγο, κάνουμε για την ευρωπαϊκή αρχή εργασίας και όχι μεταφορών. Άρα δεν αφορά μόνο τις μεταφορές. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω να επικεντρωθείτε σε αυτό το ευρύ φάσμα του τίτλου της αρχής αυτής. Δεν θεωρώ ότι είναι πλατφόρμα που όλοι θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσει, την ε, αμοιβή του προσωπικού κτλ. Δεν πιστεύω ότι θα μπορέσει αυτό να εφαρμοστεί μέσω κανονισμών ε, σε εθνικό επίπεδο. Αλλά μπορεί αυτός ο μηχανισμός να βοηθήσει σε περίπτωση ας απόσπασης εργαζομένων σε άλλες χώρες. Αυτό που περιμένουν από εμάς, λοιπόν, και αυτός πρέπει να είναι ο στόχο τη δημιουργία αυτού του οργανισμού. Να μπορέσουμε να αντιδράσουμε σε αρνητικά περιστατικά, σε περιπτώσεις καταχρήσεων, ε, σε οτιδήποτε δεν είναι σύμφωνο με το σύστημα. Όμως δεν συμφωνούμε ότι αυτή η αρχή θα πρέπει να ελέγχει τις επιχειρήσεις να μπαίνει, να εισέρχεται στους χώρους των επιχειρήσεων σαν ε, μέρος ε, δραστηριοτήτων καταπολέμησης απάτης. Άρα όλες οι λύσεις που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις, που παρέχουν πληροφορίες και που καταπολεμούν τις καταχρήσεις και που παρέχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση για τις μικρομεσαίε επιχειρήσει όλα αυτά θα πρέπει να υποστηριχθούν. Θεωρώ ότι αύριο θα έχουμε ένα ισορροπημένο έγγραφο τη Επιτροπής Μεταφορών που θα μας βοηθήσει όλους όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό, όχι μόνο στον τομέα των μεταφορών, και ότι θα καταπολεμηθεί μέσω αυτής της αρχής και η στρέβλωση του ανταγωνισμού. Γι' αυτό υποστηρίζουμε όλες τις καλές προτάσεις, τις ε, καλές συμβαστικές λύσεις. Έχω κάνει και εγώ σχετικές προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Σουσλοτοφσκή. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον συγητή και τους Χιώδης. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σε διάφορα σημεία καταφέραμε να αλλάξουμε το κείμενο, ωστόσο το ECR συνεχίζει να επικρίνει και να μην είναι ικανοποιημένο με τη δημιουργία μιας τέτοιας αρχής και με τόσο ευρείες αρμοδιότητες. Πρώτα απ' όλα, επειδή το εργατικό δίκαιο αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και επομένως καμία ευρωπαϊκή αρχή δεν μπορεί να έχει τόσο ευρείες αρμοδιότητες. Θα αντίκειτο στη συνθήκη. Εκτός εάν αποφασίσουν τα κράτη-μέλη κάτι διαφορετικό, αλλά μόνο τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που μπορούν να παίρνουν τέτοιες ε, ε, πρωτοβουλίες, να δημιουργούν μια αρχή η οποία θα έχει τη δυνατότητα να κάνει ελέγχους επιτόπιους, να υποβάλει πρόστιμα. Αυτά είναι αρμοδιότητες των κρατών μελών. Εμείς επίσης θα επιθυμούσαμε να αλλάξει η ονομασία της αρχής. Καλύτερα να ονομάζεται η υπηρεσία για τους εργαζομένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με, με, το τρόπο με, τον οποίο, με, αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο ξεκάθαρο ποιο είναι ο ρόλος της, γιατί στην πραγματικότητα παρέχει πληροφορίες για κάποιον ο οποίο θέλει να εργαστεί στο εξωτερικό, σε, σε άλλο κράτο μέλο, μπορεί να οργανώνει σεμινάρια, μπορεί να παρέχει τεχνική υποστήριξη και την ανταλλαγή πληροφοριών που χρειάζεται να γίνεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εργατικής Νομοθεσίας. Όχι όμως να λειτουργεί σαν αστυνομία ως ελεγκτικός μηχανισμός υπέρ των αποσπασμένων εργαζομένων στην Ευρώπη, όχι να μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα στις επιχειρήσεις. Επίσης, θα θέλαμε οι εργοδότε να, να, από τη δημιουργία αυτή τη αρχή. Ιδιαίτερα οι εργοδότε εκείνοι οι οποίοι υφίστανται δυσμενεί διακρίσει από τις αρχές τις εθνικές ε, αγοράς εργασίας, του ελέγχου τη αγορά εργασία του. Με αυτόν τον τρόπο οι εθνικές ε, αρχέ επιθεώρησης εργασίας δημιουργούν εμπόδια στη δημιουργία της ενίας αγοράς και μια τέτοια ευρωπαϊκή αρχή, όπως εμείς τη φανταζόμαστε, θα μπορούσε να, να βοηθήσει ώστε αυτά να αρθούν. Έρχομαι τώρα πιο συγκεκριμένα στον τομέα των μεταφορών. Θα θέλαμε να αναφερθεί συγκεκριμένα ω τομέα μεταξύ των οποίων θα μπορούσε να ε, ασχοληθεί αυτή η αρχή. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο το γεγονό ότι η Επιτροπή Μεταφορών συζητάει αυτή την ε, γνωμοδότηση. Δεν σημαίνει ότι θέλουμε να τιμωρήσουμε τους εργοδότε στον τομέα των μεταφορών. Θέλουμε να βρούμε για αυτούς λύσεις, έτσι ώστε να δραστηριοποιούνται στην νέα αγορά. Με αυτήν τη φιλοσοφία υποβάλαμε εμεί τι τροπολογίε μα. Ορισμένε από τι θέσει μα συμπεριλήφθησαν στις ε, συμβιβαστικέ. Όμω, εμεί επιμένουμε στι προτάσει μα στι υπόλοιπε που δεν μπήκαν και θα προτιμούσαμε να καταψηφιστεί και η έκθεση συνολικά. Η κυρία Βραντίκα Μπιλμπάου. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντέτσεν, τον εισηγητή, για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει και γιατί ήταν πολύ δύσκολο να συντονίσει όλες αυτές τις εργασίες. Εμείς συμφωνούμε με τους συμβιβασμούς ως ε, φιλελεύθεροι. Εάν αξίζει κανείς να είναι ευρωβουλευτής για ορισμένες εκθέσεις, αυτή είναι μία από αυτές. Έχουμε μία γνωμοδότηση για τον τομέα των μεταφορών, ο οποίος χαρακτηρίζεται από μεγάλη κινητικότητα. Δύο εκατομμύρια διαβαίνουν τα σύνορα κάθε ημέρα μεταφέροντας εμπορεύματα ή αγαθά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η πρόταση ε, θα ενισχύσει τον κοινωνικό πυλώνα και εμείς ως ε, πολιτική ομάδα καθώς και εγώ ως Ευρωβουλευτής τόνισα ότι έπρεπε να ενισχύσουμε τον κοινωνικό πυλώνα. Ήμασταν υπέρμαχοι αυτού εξ αρχής. Και στο Γκέτεμπορκ έγιναν συγκεκριμένες συστάσεις και γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Επίσης θα πρέπει να μιλάμε για το γεγονός ότι οι πολίτες ζητούν απαντήσεις. Μιλάμε για ε, μετακίνηση 2 εκατομμυρίων την ημέρα και φυσικά οι νέοι έχουν πολύ μεγαλύτερη κινητικότητα, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι μέχρι τώρα. Σε τρεις, τέσσερις ή πέντε χώρες θα πρέπει να συντονιστούν οι δράσεις των οργανισμών στα κράτη για να έχουν πληροφορίες και να βρουν λύσεις. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι ένα μέσον που μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερη Ευρώπη για να βελτιώσουμε την κατάσταση και τα δικαιώματα των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Αυτό θα ευεργετήσει τους πάντες. Ελπίζω τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν με την εφαρμογή της νομοθεσίας και να λειτουργήσει αυτός ο συντονισμός που δεν μπορεί να γίνει από μόνος του από το Ευρωκοινοβούλιο. Γι' αυτό σκεφτόμαστε τους πολίτες και πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσουμε Ευρώπη με μεγαλύτερη ευημερία. Γι' αυτό και για πολλούς άλλους λόγους υποστηρίζουμε τους 17 συμβιβασμούς που έχουν υποβληθεί και μια σειρά τροπολογιών. Η κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστούμε μάλλον κυρία Μπιλμπάου. Και εγώ είμαι σκιώδης και θα λάβω τώρα το λόγο. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα σημείο κλειδί για την εντολή και τη θητεία μας. Είναι ένα μέσον και θα ήθελα να λάβετε υπόψη ότι επειδή μιλάω να κάνετε λίγη ησυχία. Η Ευρώπη δεν είχε αυτή την εργαλειοθήκη έτσι ώστε να ορίσει τη συλλογιστική αυτή της Ευρώπης όταν μιλάμε για την κοινωνική πτυχή. Πολλές φορές χρησιμοποιούσαμε μια λέξη, το κοινωνικό dumping. Αλλά το θέμα του κοινωνικού dumping αφορά και τον τομέα των μεταφορών. Εάν σήμερα δεν μπορέσουμε να αναλύσουμε και να διαδώσουμε πληροφορίες του άμεσα εμπλεκόμενους, τότε δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Έχετε δίκιο, κυρία Μπιλπάου. Θα πρέπει να θέσουμε ενώπιον των ευθυνών του στα κράτη-μέλη. Αυτός ο οργανισμός υπάρχει για να εποπτεύει, έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι να διαθέτουν πολύ καλύτερες και υγιείς συνθήκες κάτι το οποίο βοηθάει τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους αλλά και το κοινό, το ευρύ κοινό, έτσι ώστε να προληφθούν μεγάλοι κίνδυνοι όταν μιλάμε για την εργασία, αλλά και με ένα στόχο. Όποιος και να είναι ο τομέας, θα πρέπει να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη. Ο οργανισμός αυτός θα πρέπει να συντονίσει και να προτρέχει των νομοθετικών αλλαγών που είναι σημαντικές για τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό είναι και ένα μέσο ευαισθητοποίησης, ε, κύριε εισηγητά. Γιατί πολύ συχνά όταν μιλάμε για οργανισμούς λέμε, έχουμε πληθώρα οργανισμών. Όμως αυτός ο οργανισμός είναι η κινητήριος δύναμη της κοινωνικής πτυχής. Γι' αυτό θα πρέπει και ως προς τη λειτουργία του να βοηθήσουμε όλοι έτσι ώστε να εκπονήσει στρατηγικές και στόχους που θα οριστούν έτσι ώστε αυτός ο οργανισμός να είναι λειτουργικός. Εμείς πάντα θα προβάλλουμε την θεώρηση της Επιτροπής μας και θα ε, λάβουμε υπόψη και επιμέρους ε, ζητήματα, γιατί αν δεν χτίσουμε την κοινωνική Ευρώπη, τον κοινωνικό πυλώνα, δεν τον καταφέρουμε τότε, δεν θα τον χτίσουμε ποτέ. Η κυρία Κιλόνεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, έχω μια επιστολή από την Τάνια Κονσάλες Πένιας, ε, που είναι σκιώδης μας και θα σας τη διαβάσω. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για την συνεργασία που είχαμε. Όπως όλοι γνωρίζετε, η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής που θα έχει τον στόχο την ενίσχυση των ίσων δικαιωμάτων και των ευκαιριών για τους εργαζόμενους που κινούνται διασυνοριακά εντελώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να δώσουμε ξεκάθαρες αρμοδιότητες σε αυτή την αρχή, έτσι ώστε να μπορέσει αποτελεσματικά να παίξει το ρόλο της. Γι' αυτό το λόγο θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα των συναντήσεων των σκιωδών και τις ε, συμβεβαστικές τροπολογίες. Ο Ζαν Κλοντ Ιούκερ ανέφερε με το ε, ε, ρητά ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας τέτοιος φορέας και όχι μια τέτοια υπηρεσία. Βεβαίως χρειάζεται συνεργασία με τα κράτη-μέλη θα χρειαστεί αυτή η συνεργασία για να λεφθούν οι πληροφορίες, έγγραφα. Αυτό θα είναι απαραίτητο για να μπορέσει αυτή η υπηρεσία να, να παίξει το ρόλο της. Θα χρειαστεί επίσης συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, να λαμβάνει πληροφορίες από αυτούς, έτσι ώστε να εντοπίζει που υπάρχουν προβλήματα με την ελεύθερη ε, ε, ε άσκηση των εργατικών δικαιωμάτων ή παρατυπίες στην αγορά εργασίας. Γνωρίζουμε ότι τέτοιες πρακτικές μπορεί να ε, εφαρμόζονται σε διάφορες σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους εργαζόμενους που εργάζονται διασυνοριακά. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η αρχή να συλλέγει και να δημοσιοποιεί ακριβείς πληροφορίες για το εργατικό δίκαιο σε όλες τις γλώσσες και να δημοσιοποιεί αυτές τις πληροφορίες με τρόπο εύχριστο προς το χρήστη. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να φροντίσουμε επιτέλους τα δικαιώματα εκείνων που εργάζονται στο εξωτερικό, σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να οικοδομήσουμε την κοινωνική Ευρώπη, δίνοντας εργαλεία στους πολίτες μας, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν ικανοποίηση από την εργασία του χωρί να υφασίσταν διακρίσει όπου και αν βρίσκονται στο εσωτερικό τη Ένωση. Ελπίζω αύριο στην ψηφοφορία να εγκρίνουμε μια φιλόδοξη τέτοια εντολή, να ζητήσουμε να δημιουργηθεί μια τέτοια αρχή. Αυτό θα βοηθήσει ιδιαίτερα τον τομέα των μεταφορών, έναν τομέα στον οποίο ε, σημειώνονται σημαντικέ παραβιάσει όσον αφορά το εργατικό δίκαιο. Σα ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη. Σα ευχαριστούμε κυρία Κίλωνα και κυρία Γεβονταλώνη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Από τη συνάδελφη, το είχα πει και κατά την παρουσίαση της επιτρο... Ε, έκθεσης, η δημιουργία μια τέτοια αρχή είναι κάτι που χρειάζεται εδώ και πολύ καιρό. Χρειάζεται, το ζητάει εδώ και πολύ καιρό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι απαραίτητο να έχουμε μια αρχή που θα φροντίζει για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού ε, εργατικού δικαίου. Έχουμε αντίστοιχες αρχές ε, για να εφαρμόζεται, για παράδειγμα, το δίκαιο ανταγωνισμού σε ολόκληρη την νέα αγορά. Γιατί όχι, λοιπόν, και μια αντίστοιχη αρχή για να εγγυάται τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων. Θα ήθελα να χαιρετήσω το εξαιρετικό έργο που έκανε ο εισηγητής μας. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω σε όλου του αδελφού να μην ψάξουμε τον ελάχιστο κοινό να μην δημιουργήσουμε μια αρχή η οποία απλώ να βοηθάει με πληροφορίε τι εθνικέ αρχέ. Πρέπει να τη δώσουμε την αρμοδιότητα να κάνει ελέγχου και, εάν χρειάζεται, να επιβλέπει και τι εθνικέ αρμόδιε αρχέ. Σα ευχαριστούμε, κυρία Γαβενταλόν. Κύριε Φανερκάμπ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ενδιαφέρον ότι πήρα το λόγο με τον προηγούμενο μιλητή, γιατί έχω τελείως διαφορετική άποψη. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους σκιώδες εισηγητές, αλλά πρέπει να δούμε τι διακυβεύεται εδώ. Η κοινωνική πολιτική ε, αφορά τα κράτη-μέλη. Κάθε κρατός μέλος έχει διαφορετικό κοινωνικό σύστημα και αυτά τα συστήματα δεν είναι συμβατά. Ίσως στο μέλλον το βιωτικό επίπεδο στη Ρουμανία να είναι το ίδιο στο επίπεδο με αυτό στην Ολλανδία. Όμως αυτό δεν συμβαίνει τώρα και θεωρώ ότι, ότι προχωράμε, τραβάμε λίγο το σκηνή όσον αφορά τις εθνικές ε, αρμοδιότητες γιατί οι θα μπορούν να ασκήσουν το έργο τους καθώς η Ευρώπη θα το αναλάβει. Όπως τον οδικό κλάδο, παραδείγματος χάρη, αν δούμε υπάρχει τουρισμός ε, διασυνοριακός, δεν υπάρχουν κίτρινα. Ουσιαστικά αυτό που κάνετε είναι να αναλαμβάνετε εσείς τις εθνικές αρμοδιότητες. Δείτε την έκθεση και θα δείτε ποια θα είναι η λειτουργία της αρχής σε σχέση με τις εθνικές επιχειρήσεις. Δεν το συντονίζεται. Ουσιαστικά μεταφέρει όλες τις αρμοδιότητες στην, Εθνική Αρχή, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Θεωρώ όμως ότι τραβάμε το σκηνή όσον αφορά την κοινωνική πολιτική. Έτσι όμως δεν ενισχύεται τον κοινωνικό παράγοντα. Και αυτό είναι κάτι με το οποίο συμφώνησε η κυρία Λουιτσέσκα. Ευχαριστώ κύριε Γκάμπ. Η κυρία Γκραπίνη. Ευχαριστώ. Ξεκινώ από την ιδέα ότι και η χώρα μου και εγώ συμφωνήσαμε με την πρόταση της Επιτροπής να υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας όχι μόνο για τις μεταφορές, αλλά και για τις ε, μεταφορές. Ε. Πρόκειται για μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας γενικότερα, όπως ορίζει και ο τίτλος. Ο κύριος Βαντεκάμπ ανέφερε, για, αναφέρθηκε στις τροπολογίες μου. Αυτή η πλατφόρμα, αυτή η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας είναι μια πλατφόρμα η οποία συνδέει τις εθνικές αρχές μεταξύ τους έτσι ώστε να γίνεται διαβίβαση ευκολότερα των πληροφοριών, έτσι ώστε ο πολίτης να τις ε, ε, διαθέτει. Αν εγώ ως ΜΜΕ θέλω να ε, μεταβώ σε μία άλλη χώρα, δεν ξέρω πώς έχει η εργασία εκεί, πώς ορίζεται ένα πλαίσιο εργασίας. Γι' αυτό χρειάζεται αυτή η πλατφόρμα. Φυσικά, η Επιτροπή είπε ότι θέλουμε να αυξήσουμε την ισότητα στην αγορά εργασίας. Όλοι θέλουμε την ισότητα. Εγώ ε, προέρχομαι από μία χώρα της Ανατολικής Ευρώπης και είναι πολύ δύσκολο να ανταγωνιστούμε τις μεγάλες εταιρείες της δύση. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει εξισορρόπηση μεταξύ επικουρικότητας και του τι μπορεί να γίνει με αυτή την αρχή. Εγώ υπέβαλα μία τροπολογία με μία συμπλήρωση, ένα συμπλήρωμα σε σχέση δηλαδή με την εποπτεία και τους ελέγχους. Θα πρέπει να γίνονται εθνικές επιθεωρήσεις. Δεν μπορεί κανείς να βραχικυκλώσει το όλο σύστημα. Πρέπει να έχουμε όλα τα στοιχεία και αυτό θα πρέπει να γίνει με βάση τις εθνικές αρχές. Γιατί αν έρθει κάποιος ε, στην Ρουμανία να επιθεωρήσει και βασιστεί στο γερμανικό νόμο ή στον Ολλανδικό, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό θα πρέπει να αξιολογήσουμε τους κινδύνους. Εάν γίνει η αποτίμηση κινδύνων, θα πρέπει να βασιστούμε σε όλα τα κράτη-μέλη. Έχω και μία τροπολογία που δεν ξέρω κατά πόσο θα περάσει. Εδώ στην έκθεση υπάρχει και το θέμα της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα μπορούσαν όλοι να είναι Ολλανδοί ή Γερμανοί. Νομίζω θα πρέπει να υπάρχει και ένας γεωγραφικός επιμερισμός γιατί οι αγορές εργασίες έχουν, εργασίες έχουν ιδιαιτερότητες. Η αρχή αυτή θα πρέπει να ε, προβάλλει στοιχεία και επιγραμμικά και online για να δούμε κατά πόσο υπάρχουν ε, προβλήματα στην λειτουργικότητα και για να μην υπάρχουν δυσλειτουργίες. Ελπίζω να ρυθμίσουμε το όλο πλαίσιο, διαφορετικά δεν θα έχουμε καταφέρει τίποτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Ντέτχεν για, για το έργο σας. Σας άκουσα με προσοχή. Κάνετε λόγο για τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας και έτσι όπως ε, το αποτυπώσετε, είναι σαν να μιλήσετε για μια αρχή που θα ασκεί ελέγχου οδικούς. Έχει να κάνει με την κινητικότητα των εργαζομένων και να την προωθήσει και όχι να ορίσει τις διατάξεις και τις προδιαγραφές ε, για τον τομέα των μεταφορών. Αυτό είναι γιατί πρέπει να προσέξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup, Monsieur Σας ευχαριστώ, κύριε Ντεμόντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι υπέρ της θέσπισης αυτής της αρχής και χαίρομαι γιατί μιλάμε για αρχή, όπως είπε και κάποιος ε, προλαλή σας. Αυτή η αρχή διαδρά με την εσωτερική αγορά για την ελευθερία εγκατάστασης, μεταφορά αγαθών και εμπορευμάτων και θα πρέπει να υπάρχει μία δίκαιη ε, ρύθμιση και ένα δίκαιο κανονιστικό πλαίσιο στα κράτη-μέλη για να καταπολεμηθούν οι καταχρήσεις και να υπάρχει καλύτερη εφαρμογή των χρηστών πρακτικών. Ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο εκατομμύρια εργαζόμενοι που ε, αλλάζουν, που περνούν τα σύνορα κάθε μέρα και υπάρχουν πολλά ε, αρνητικά στοιχεία σε αυτές τις ε, διελεύσεις. Γι' αυτό χρειάζονται πιο σαφείς ε, ρυθμίσεις. Εγώ θεωρώ ότι ως Επιτροπή δεν βελτιώσαμε το ρυθμιστικό πλαίσιο γιατί αν μιλάμε για ψηφιοποίηση, αν μιλάμε για κανονιστικό πλαίσιο βελτίωσης των συνθήκων εργασίας των εργαζομένων, θα πρέπει να έχουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο ως βάση. Διαφορετικά στην ουσία φτιάχνουμε, ορίζουμε μόνο το τελευταίο, την τελευταία ψηφίδα, ενώ δεν υπάρχουν οι οι βάσεις. Βαντάλεν. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, είναι προφανές ότι υπάρχουν προβλήματα στον τομέα των μεταφορών, των οδικών μεταφορών ιδιαίτερα. Δεν υπάρχει ίση αμοιβή για ίση εργασία. Υπάρχουν διαφορέ ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη κάνουν τι επιθεωρήσει και του ελέγχου των οχημάτων και των οδηγών και θα μπορούσα να αναφέρω και πολλά περισσότερα προβλήματα. Όμως εδώ έχουμε μια κλασική αντίδραση του σκυλιού του Παυλόφ από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το που ακούει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, να λύξουμε το πρόβλημα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ως συνήθως γίνεται μια επίκληση του συντονισμού Αλλά αυτό κατά την άποψή μου είναι προσχηματικό. Είναι αυτό που πάντα αναφέρουμε όταν θέλουμε να ε, λύσουμε ένα πρόβλημα που δεν ξέρουμε πώς να το λύσουμε, τι λέμε, να δημιουργήσουμε και ακόμα μερικές αρχές που θα κάνουν ακόμα περισσότερους ελέγχους, ας βάλουμε και ορισμένες άλλους να ασχοληθούν δηλαδή. Στην πραγματικότητα όμω, όπω είπε και μια συνάδελφο πριν, αυτό απλώ θα δημιουργήσει ένα βραχυκύκλωμα. Θα ε, εξευτελιστούμε αν θέλετε, γιατί για άλλη μια φορά θα δουν οι πολίτε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να του βοηθήσει ακριβώ εκεί που είναι ε, τα πραγματικά του καθημερινά προβλήματα. Τι θα καταφέρουμε, απλώ θα δημιουργήσουμε ακόμα μια υπηρεσία με τη γραφειοκρατία τη. Χωρί να αλλάξει κάτι. Άκουσα συναδέλφου που πιστεύουν ότι αυτό είναι, θα ήταν ένα θετικό βήμα, ότι θα βοηθήσει και του τους πολίτες, ότι θα βοηθήσει και τις επιχειρήσεις, ότι θα βοηθήσει τον συντονισμό. Αλλά εμένα μου φαίνεται ότι απλώ έχουμε ένα πρόβλημα και του πετάμε ε, χρήματα ελπίζοντα ότι θα φτιάξει. Δεν πιστεύω ότι γίνονται έτσι τα πράγματα. Σα ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο και στον κύριο Ζεντό από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόληση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την μας εκθέσει και τη θέση της ε, Επιτροπής. Πράγματι, ονομάζομαι Ζοντό. Δεν συνηθίζεται να, να εκπροσωπώ την Επιτροπή στην Επιτροπή Μεταφορών. Σε ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την ε, ευκαιρία που μου δίνετε. Σας ευχαριστώ επίσης και τον εισηγητή σας και όλους για το έργο σας. Υποστηρίζουμε αυτή την πρόταση. Την είχαμε υποβάλει το Μάρτιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ό,τι, γίνει, ό,τι μπορεί για να εγκριθεί η δημιουργία αυτής της αρχής μέχρι το τέλος της θητείας. Συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλες τις άλλες συναρμόδιες επιτροπές και φυσικά συνεργαζόμαστε και με το Συμβούλιο. Είχαμε λοιπόν πολλές και διάφορες συζητήσεις. Έχουμε ακούσει πολλές και διαφορετικές θέσεις, απορίες, ανησυχίες, παρατηρήσεις σε σχέση με την επικουρικότητα, σε σχέση με τις αρμοδιότητες που θα έχει αυτή η αρχή και ακόμα και αυτό που λέγεται ότι απλώς δημιουργούμε ακόμα μια γραφειοκρατική αρχή. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι οι αρμοδιότητες που προτείνει, προτείνονται για αυτή την αρχή είναι αρμοδιότητες που ήδη υφίστανται. Ορισμένες ήδη προβλέπονται μερικώς στην νομοθεσία και άλλες είναι καινούργιε. Επομένω, αυτό που προτείνουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να συνεχιστεί αυτό που λειτουργεί και να προσθέσουμε σταδιακά και κάποια ακόμα στοιχεία. Γιατί, γιατί έχουμε μια, ένα τομέα στον οποίο πρέπει να συνεργαστούμε περισσότερο στενά. Και ο στόχος είναι να προωθήσουμε την κοινωνική ασφάλεια, το, το, τους, τα δικαιώματα των εργαζομένων και την κινητικότητα. Έρχομαι λοιπόν στο ζήτημα τη κινητικότητα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και γνωρίζουμε ότι η κινητικότητα αυξάνεται κάθε χρόνο. Έχουμε και όλο και περισσότερου εργαζόμενου που εργάζονται σε κάποιο άλλο κράτο μέλο. Επομένω, δεν χρειάζεται να κάνει κανεί διαφήμιση. Η κινητικότητα των εργαζομένων αυξάνεται από μόνη τη. Όμω, οι ενδιαφερόμενοι, είτε αυτοί είναι οι δημόσιε αρχέ, είτε είναι οι επιχειρήσει, είτε είναι οι εργαζόμενοι, θα πρέπει να έχουν στα χέρια του ένα εργαλείο που θα τους δώσει τη δυνατότητα να έχουν καλύτερες πληροφορίες στη διάθεσή τους, να μπορούν να συνεργάζονται καλύτερα και σε ορισμένες περιπτώσεις αυτή η αρχή να κάνει και προτάσεις για βελτίωση και για λύσεις. Αυτές είναι λοιπόν οι βασικές αρμοδιότητες. Συλλογή πληροφοριών και ενημέρωση, συνεργασία και διαμεσολάβηση. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, προσοχή που δόξατε στο θέμα. Συνεργαζόμαστε και με την Επιτροπή ε, Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι ώστε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας ε, της ε, διαδικασία δηλαδή των τριμερών διαλόγων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ. Και εμεί σα ευχαριστούμε κύριε Ζωντώ. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μα. Ja, vielen Dank. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ούτε καμιλές βλέπω, ούτε συνέλευση το πανηγυρίζουν. Θεωρώ ε, με τον κόνοπα και καταπίνουμε την κάμιλο με αυτή την έκθεση. Είναι μια ισορροπημένη έκθεση όσον αφορά και την επικουρικότητα και την οπτική που έχει η Επιτροπή Μεταφορών. Κύριε Βάντερ Κάμπ, δεν έχει να κάνει με το να κλέψουμε αρμοδιότητες από τις εθνικές αρχές, αλλά να τις υποστηρίξουμε στο έργο τους. Και αυτό φαίνεται στην έκθεση. Έχει να κάνει με τη συγκέντρωση πληροφοριών, την απλούστευση των διαδικασιών, προς όφελος των πολιτών και προς όφελος των συστημάτων, των κοινωνικών συστημάτων. Ευχαριστώ πολύ. Αύριο θα το συζητήσουμε και περισσότερο. Θα ψηφίσουμε αύριο στις 9 το πρωί. Και συνεχίζουμε. με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές διεξουδίου του άνθρακα των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Η κυρία Βερκούνεν έχει το λόγο. Yes, thank you, Madam Chairman. Um, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι ένας πολύ σημαντικός κανονισμός. Θα δώσουμε την γνωμοδότησή μας στην Επιτροπή ε, Περιβάλλοντος, που είναι επί της ουσίας Επιτροπή την προηγούμενη φορά στην Ολομέλεια κάναμε λόγο ψήφισμα για τα οχήματα. Είχαμε δυσκολίες να πετύχουμε πλειοψηφία και σύμφωνη γνώμη εντό των πολιτικών ομάδων. Ελπίζω ότι θα είναι πιο εύκολο με αυτό το φάκελο. Γνωρίζουμε ότι είναι μια, ένας πολύ σημαντικός κανονισμός και η Επιτροπή προτείνει τους ίδιους στόχους για τα ε, βαρύ επαγγελματικά οχήματα όπως και για τα επιβατικά 50% ως το 2025 και ως το 2030. Even that this is first time when we... Υψηλότερο ποσοστό. Θέτουμε στόχους ε, για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, οι οποίοι γνωρίζουμε ότι είναι πολύ αποτελεσματικοί γιατί η κατανάλωση καυσίμων ίσως είναι το πιο σημαντικό θέμα όταν αγοράζουμε βαρέα οχήματα, γιατί κανείς δεν οδηγεί προς ε, για να διασκεδάσουμε αυτά τα οχήματα είναι για εργασιακού καθαρά λόγους και άρα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αποδοτικότητα γιατί είναι πολύ ακριβά τα καύσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό τα επαγγελματικά οχήματα συνήθω είναι αποδοτικά και συνήθω μπορούμε να ε, συμφωνήσουμε με τι ε, ομάδε που θα υποστηρίξουν την πρόταση τη Επιτροπή για το 50% στο 2025 και 30% ως το 2030. Είναι μια πρόκληση και ένα φιλόδοξο σχέδιο, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι οι κατασκευαστές προσπαθούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Έχουμε 162 τροπολογίες και προτάσεις προς τις δύο κατευθύνσεις για το πόσο φιλόδοξοι είναι η στόχη που θέτουμε, αλλά μετά από συζήτηση κατανοήσαμε ότι οι πιο πολλές ε, πολιτικές ομάδες είναι πρόθυμες να υποστηρίξουν την πρόταση της Επιτροπής. Οι υπόλοιπε τροπολογίε ε, εστιάζουν σε μεθόδους υπολογισμού. Υπήρξαν πολύ καλές προτάσεις για τους υπολογισμούς και τώρα και στο μέλλον. Επίσης, προετοιμάζουμε τη συμβαστική 8 όταν θα εκδώσει την έκθεση της Επιτροπή το 2022 θα πρέπει σε αυτό το χρονικό πλαίσιο ε, να κάνουμε λόγο για τις μετρήσεις από φρέαρ στον τροχό και τον κύκλο των εκπομπών. Άρα αναμένουμε ότι η Επιτροπή θα εργαστεί πιο δυτικά σε αυτό το πεδίο γιατί δεν είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το σύστημα υπολογισμών όπως ε, ισχύει ως τώρα. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω με βάση την κατανάλωση από φρέαρ στον τροχό. Από εδώ και στο εξή. Έχουμε λοιπόν 162 τροπολογίες και σχεδιάζουμε 12 συμβαστικές ήταν πολύ δραστηρικές και οδησίτες. Θέλω να του ευχαριστήσω όλους και ελπίζω ότι μπορούμε να την εγκρίνουμε την ε, γνωμοδότηση αύριο, ώστε να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στην Επιτροπή ε, Περιβάλλοντος που είναι η Επιτροπή. Επιτροπή. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, Madame κυρία Βιρκούνεν. Η κυρία Ρεβονταλόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Η έκθεση ε, είχε απήχηση στον ε, τύπο. Φυσικά μιλάμε για μείωση του, των εκπομπών διοσιδίου του άνθρακα και μιλάμε για ανάγκη για, ώστε να υπάρχουν πρότυπα μέχρι το 2025 είτε για τα ελαφρά είτε για τα βαρέα οχήματα. Γι' αυτό θα γίνει μία αναθεώρηση το 2022 γιατί δεν μπορούμε να ορίσουμε τις προθεσμίες σωστά. Για κάθε υπομάδα οχημάτων θα πρέπει να ορίσουμε συγκεκριμένα όρια, κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό χαίρομαι που όλοι θα συμμετάσχετε σε αυτό το λογισμικό και στην κατάρτισή του. Όμως αν θέλουμε ε, να αλλάξουμε τα πλαίσια για τις μηδενικές ή απειροελάχιστες εκπομπές, στην ουσία ε, μετράμε τα οχήματα επί 2, 3 και 4. Και γι' αυτό νομίζω ότι δεν γίνονται ουσιαστικές μειώσεις, αλλά ε, απλώς δίνουμε ένα πλαίσιο και χτενίζουμε το κείμενο. Τώρα, σε σχέση με τα οχήματα μηδενικών εκπομπών και για την ε, τεχνολογική ουδετερότητα συμφωνούμε, αλλά θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε ε, πολύ σε σχέση με τις μηδενικές εκπομπές ή τις απειροελάχιστες ε, εκπομπές και τις υπερπιστώσεις όπως ορίζονται. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντεμασμέκερ θα λάβει το λόγο εξ ονόματος του κυρίου Ζήλενε ναι ή όχι. Όχι. Όχι. Εντάξει. Ο κύριος Ράντος. Thank you very much. Uh, I, I would like to thank... Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή και τους συναδέλφους Σκιώδης για την καλή συνεργασία που είχαμε. Η Άλντε υποστηρίζει την έκθεση, υποστηρίζει και τον κανονισμό. Όσον αφορά τα, τις προτάσεις της Επιτροπής για τα επιβατικά, Νομίζω ότι και, αυτά, και αυτές είναι αρκετά φιλόδοξες. Βεβαίω χρειάζεται να αναθεωρηθεί ο κανονισμός για να αλλάξει η μεθοδολογία του υπολογισμού. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε φορά αλλάζουμε τους στόχους μας, κάθε φορά που συζητούμε δηλαδή το θέμα, και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στις επιχειρήσεις, στην αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία πρέπει να ακολουθεί αυτέ τι αλλαγές και κάθε φορά να προσαρμόζεται. Θα δούμε όμως πώς θα εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα και πού θα οδηγήσει τελικά αυτός ο κανονισμός. Σας ευχαριστώ. Merci beaucoup, monsieur Ευχαριστούμε, κύριε Αντός, κύριε Το 1 τέταρτο των συνόλου των εκπομπών από τον τομέα των μεταφορών προέρχεται από τα βαρέα οχήματα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να θέσουμε φιλόδοξους νέους κανόνες για αυτά τα οχήματα και να εφαρμοστούν. Καλωσορίζουμε λοιπόν το γεγονό ότι συζητιέται αυτή, αυτό το θέμα στην Επιτροπή. Ωστόσο, αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι έχουμε ξεχάσει στις συμβιβαστικές λύσεις και συμφωνίες ε, τους στόχους του κλίματος. Θεωρούμε ότι αυτή η μείωση κατά 30%, 30 στο 2030 είναι ε, ανεπαρκής για να πιάσουμε τους στόχους των Παρισίων. Θα έπρεπε να θέσουμε πιο φιλόδοξους στόχους γιατί όλοι επηρεαζόμαστε από αυτά τα βαρέα οχήματα. Η δικιά μας πρόταση ήταν μείωση κατά 50% και αυτό είναι κατά τη γνώμη μας απαραίτητο. Η μείωση των εκπομπών ε, μακροπρόθεσμα είναι καλύτερο και για την αυτοκινητοβιομηχανία. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουν μεγαλύτερη βεβαιότητα οι αυτοκινητοβιομηχανίες και θα φτιάχνουν πιο αποτελεσματικά αυτοκίνητα και αυτό θα αυξήσει και την ανταγωνιστικότητά τους. Υπάρχουν πολλά παραθυράκια στην νομοθεσία και οι πράσινοι είναι ιδιαίτερα, ε, ανησυχούν ιδιαίτερα για τις υπερπιστώσεις. Αυτό μπορεί σοβαρά να υπονομεύσει τη δυνατότητά μας να πιάσουμε τους στόχους μας. Με λίγα λόγια λοιπόν θεωρούμε ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να προωθηθεί πολύ πιο περισσότερο, να θέσουμε πολύ πιο φιλόδοξους στόχους, εάν είναι να πιάσουμε τους στόχους που θέσαμε στο Παρίσι. Κύριε να έχετε το λόγο. Έχω και πάλι μια επιστολή από την Γκοζάλης Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους ηγητές, τους και ηγητές για τη συνεργασία. Θα ήθελα να επιστρέψω την προσοχή σας στην έκθεση του, της ομάδας των του IPCC. Χθες λοιπόν σε αυτή την έκθεση 90 επιστήμονες από πολλές χώρες κάλεσαν τις κυβερνήσεις ε, όλου του κόσμου να δώσουν στη ηχεία για τις ε, εκπομπές οι οποίες θα πρέπει να μειθούν κατά 15% μέσα στα επόμενα 10 χρόνια γιατί κατάλαβαν ότι ο περιορισμός της πεθέρμας του πλανήτη κατά 1,5 βαθμούς είναι κάτι που πρέπει να γίνει αναγκαίο και είναι απαραίτητο γιατί τα επιδράσεις είναι μη αναστρέψιμες και για τους ανθρώπους και για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και τη ζωή στον πλανήτη. Οι επιδράσει θα είναι καταστροφικές αν δεν το καταφέρουμε αυτό Πιστευόμαστε αυτή την έκθεση και τονίζει αυτή η έκθεση ε, το τέλος της εποχής των ορυκτών καυσίμων. μέχρι το 2030 στόχο πρέπει να είναι το 45% της μείωσης και μέχρι το 2050 το 50%, 2040 το 50%. Τα αποτελέσματα των συνεδριάσεων με τους κοιόδες συνεγητές δεν καταφέραμε να πετύχουμε φιλόδοξες, φιλόδοξους στόχους, να θέσουμε φιλόδοξους στόχους αυτό που προτείνεται για την μείωση κατά 30% ε, στο 2030 δεν είναι επαρκές. Μας φαίνεται αστείο. Γιατί χαμηλή εκπομπής ε, οχήματα θα πρέπει να πετυχαίνουν τους στόχους. Αν παραμείνουμε σε αυτή τη θέση, εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμυρίων θα πληγούν από τις αυξημένες θερμοκρασίες, από τις εκπομπές, θα εκτεθούν σε ε, νοσήματα εξαιτίας ε, των κουνουπιών που θα μετακινηθούν σε άλλες περιοχές, ε, σε όλες τις υπήρους θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε κατά δύο το άτομο, τα, τον αριθμό των ατόμων που εκτίθενται σε αυτές τις συνθήκες και επίσης η έκθεση κρούει το συναγερμό για τις χώρες της Μεσογείου. Υποστηρίζουμε τις περισσότερες συμφιβαστικές και καλούμε και την υπόλοι... τις ομάδες να σκεφτούν τις επιπλοκές του να παραμείνουμε στα χαμηλά ποσοστά. Γιατί αν γίνει κάτι τέτοιο, η ευρυνή ψηφορία θα είναι μια μέρα την οποία θα μετανιώνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Κιλόνεν. Έχετε δίκιο. Απόλυτο. Όλα αυτά που περιγράψατε, γιατί δείχνουν πόσο επίγον είναι το θέμα. Να παραμένουμε άπραγοι ακόμα μπροστά στην κλιματική αλλαγή είναι ασυγχώρητο, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι ασυγχώρητο γιατί όλοι γνωρίζουμε, όλοι έχουμε τα στοιχεία στα χέρια μας. Φτάνουν πια τα συνέδρια, οι συζητήσεις. Ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση, γρήγορα. Τώρα. Αυτή λοιπόν η μετάβαση σε μια πιο φιλική προς το περιβάλλον οικονομία που συζητάμε τόσο καιρό δεν έχει ακόμα συμβεί στον τομέα των μεταφερών, που είναι ο τομέας ο οποίος ε, έχει τη μερίδα του λέοντος από την πλευρά της εκπομπής αερίων ε, του θερμοκηπίου, το 20%. Το 60% του διοξιδίου του άνθρακα προέρχεται τις μεταφορές, το 20% του συνόλου. Και τι κάνουμε, Έχουμε την έκθεση της κυρίας Βίρκουναν και θα πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Εμείς εδώ από την Επιτροπή των Μεταφορών που είμαστε φιλόδοξοι για να μην επαναληφθούν αυτά που είδαμε στην Ολομέλεια την προηγούμενη εβδομάδα. Χρειάζεται να δείξουμε τη σημασία των οδικών μεταφορών για την προστασία του κλίματος, γιατί αυτό που δεν έχει συμβεί ακόμα είναι πλέον απολύτως απαραίτητο να συμβεί για την, για την επιβίωση της ανθρωπότητας. Κυρία Βέρκουναν, λοιπόν, ελπίζω ότι η Επιτροπή Μεταφορών αύριο θα έχει και το θάρρος να, και, και, την πολιτική βούληση να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα όχι μόνο προς το σύνολο του υπολείπου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά επίσης και στους αρχηγούς των κρατών, των κυβερνήσεων για να κάνουμε αυτό που πρέπει να μην συνεχίσουμε να σφυρίζουμε αδιάφοροι μπροστά σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε τον κύριο Αλεξ Πάκο Καλώ ήρθατε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί κατάφερε να οδηγήσει σε μία σύγκληση απόψεων και θα ήθελα να τονίσω την σημασία του να εγκριθεί αυτός ο κανονισμός ο τομέας αυτός δεν έχει ρυθμιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί το 6% όμως των συνολικών εκπομπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εάν δεν υπάρξει δράση, μέχρι το 2030 θα υπάρξει αύξηση 10%. Γι' αυτό υπάρχει ανάγκη δράσης για λόγους κλιματικών αλλαγών έχουμε δεσμευτεί από τη Συνθήκη των Παρισίων και θα πρέπει να εφαρμόσουμε. Ε, αυτό αφορά και τις ΜΜΕ του τομέα μεταφόρων. Έτσι εξοικονομούμε ε, χρήματα, πολλά χρήματα. Και θα πρέπει να κρατήσουμε την τεχνολογική ηγεσία μας έτσι ώστε να είμαστε στην εμπροστοφυλακή της καινοτομίας. Γι' αυτό η Επιτροπή υπέβαλε αυτή την πρόταση δύο μήνες πριν που θεωρούμε ότι είναι φιλόδοξη και ρεαλιστική. Έχει δεσμευτικό στόχο για, μέχρι το 2025 και έναν ε, στόχο για το 2030 που τον βολιδοσκοπούμε. Γιατί υπάρχουν πολύ άγνωστοι παράγοντες, γιατί είναι η πρώτη φορά που ρυθμίζουμε αυτό το τομέα με την αναθεώρηση, λοιπόν το 2022 θα έχουμε δεσμευτικούς ε, στόχους μέχρι το 2030, αλλά και θα διευρύνουμε την εμβέλεια αυτού του κανονισμού. Ευχαριστώ πολύ για την ε, σκληρή εργασία σας και προσμένουμε να συνεχίσουμε τις συζητήσεις ως συνομοθέτες. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πάκο, η κυρία Βιρκίνεν έχει το λόγο για να συνοψίσει. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω. Νομίζω ότι ακούσαμε τις ε, διαφορετικές απόψεις και όλοι τονίζουν τη σημασία ρυθμιστικού πλαισίου. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο και θα επανέλθουμε αργότερα το 2022, γιατί είναι η πρώτη φορά που γίνεται και όπως είπε και η Επιτροπή δεν έχουμε όλες τις ε, πληροφορίες για να προγραμματίσουμε το μέλλον. Όμως θα εγκρίνουμε αύριο τη γνωμοδότηση και θα συνεχίσουμε την τη συνεργασία μας με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Βερκίνεν. Θα ψηφίσουμε αύριο στις 9 το πρωί. Και όπως είπαμε, επειδή ο κύριος Σαλίνη θα φτάσει στις 4.30, διακόπτουμε για 12 λεπτά.

Mes chers collègues, nous allons reprendre notre séance. Λοιπόν, αρχίζουμε και πάλι. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Όπως σας είπα προηγουμένως, θα αρχίσουμε με την έκθεση του κυρίου Σαλίνη πριν από την έκθεση Τέλισκα. ήρθατε κύριε Τέλισκα. Α, τότε δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τη σειρά. Χωρίς μικρόφωνο η πρόεδρος. Ωραία. Ας αρχίσουμε με τον κύριο Σαλίνη, γιατί δεν έχουν έρθει ακόμα όλοι οι σκιώδεις. Καλημέρα σας κύριε Σαλίνη. Έχετε το λόγο για το διαστημικό πρόγραμμα της Ένωσης και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα. Είναι σχέδιο γνωμοδότησης της ΣΥΤΡΕ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Η εργασία αυτή για το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα έχει εξελιχθεί πολύ ικανοποιητικά. Έχουμε 270 τροπολογίες περίπου, το οποίο δείχνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εξ αρχής. Οι 270 είναι το ίμιση περίπου των 550 της Ήτρε. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι η διακυβέρνηση και η σχέση μεταξύ των τριών θεμάτων που σχετίζονται με την διακυβέρνηση της διαστημικής στρατηγικής. Προσπαθήσαμε να ορίσουμε τις αντίστοιχες αρμοδιότητες. Η ε, Επιτροπή, η CSA, που θα είναι ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διάστημα και η ΕΖΑ. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από αυτή την εργασία, διότι θέλουμε να αποφύγουμε επαναλήψεις και επικαλύψεις που δεν βοηθάν τη διακυβέρνηση και αυξάνουν και τις δαπάνες ως προς τον προϋπολογισμό Μαζί με τους συναδέλφους ε, έχουμε προβάλει μια γενική κατευθυντήρια γραμμή που να είναι σχετική με την πρόταση της Επιτροπής, ε, δηλαδή έχουν γίνει ορισμένες μικροτροποποιήσεις αλλά πρόκειται για μικρές ποσοστιαίες αναλογίες, δηλαδή το, το γενικό επιχείρημα είναι να υπάρχει εσωτερική ευελιξία, γνωρίζοντας βεβαίως ότι υπάρχει μία πρόταση για τον Γαλιλαίο και τον Κοπέρνικο που έχουν ε, ένα υψηλότερο ποσοστό και το άλλο θέμα που μας απασχολεί είναι ο περιορισμένος προϋπολογισμός ε, GovSatcom και SSA. Η πρότασή μου είναι να αυξήσουμε, να διπλασιάσουμε αν θέλετε, τα 500 εκατομμύρια που προορίζονται σε αυτά τα δύο προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό θα οδηγούσε σε μία αύξηση των επιπλέον 16 δις σε 16,7 με ορισμένες διακυμάνσεις. Και αυτό θα μας επιτρέψει αυτά τα προγράμματα να είναι λειτουργικά. Διαφορετικά στην ουσία ε, σκοτώνουμε αυτά τα προγράμματα εκγενετής. Θέλουμε λοιπόν να παγιωθούν αυτά τα προγράμματα. Δηλαδή το Γαλιλαίο και Έγνος και ο Κοπέρνικος. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σαλίνη για αυτά τα εισαγωγικά σχόλια που είναι απόλυτα σαφή. Υπάρχει πραγματική θέληση να ε, υπερασπιστούμε το διαστημικό μας πρόγραμμα για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και σε διεθνές επίπεδο. Ο κύριος Ασής. Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο ο κύριος Ασής. Το μικρόφωνο σας. Το στίχημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο διαστομικό πρόγραμμα, ιδιαίτερα για την έρευνα και την κοινοτομία, ε, είναι ένα συνενετικό πρόγραμμα και πρωταρχικός μας στόχος. Η Επιτροπή θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να είναι στην εμπροστοφυλακή του διαστήματος και θα πρέπει να εξεύρει τους πόρους τη στιγμή που χρειάζεται περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη, έτσι ώστε να έχουμε ανταπόδοση στο μέλλον. Γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να πάμε πιο μακριά είτε ως προς τα προγράμματα που προϋπάρχουν, είτε στην ε, επαναξιολόγηση των ε, μελλοντικών. Θα πρέπει λοιπόν όλες οι πολιτικές δυνάμεις να ξεκινήσουν ένα πολιτικό διάλογο. Ο εισηγητής θα τύχει της υποστήριξής μας και θα ε, ήθελα να λάβετε υπόψη τις τροπολογίες δημοσιονομικού χαρακτήρα. Υπάρχουν και πολλές τροπολογίες ε, δικές μας που δεν εντάχθηκαν στις προτάσεις συμβιβασμού, ιδιαίτερα ως προς τη βιωσιμότητα και το περιβάλλον. Είμαι σίγουρος ότι αύριο θα έχουμε να κάνουμε με μια πολύ καλύτερη πρόταση από αυτή που υπέβαλε η Κομισιόν. Έγινε συζήτηση και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Γι' αυτό θα θέλαμε να μας υποστηρίξετε στις προτάσεις δημοσιονομικού χαρακτήρα, στις τροπολογίες, γιατί είναι πιο φιλόδοξες με βάση τις προτεραιότητές μας, ιδιαίτερα σε σχέση με το τομέα των μεταφορών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Κύριε Σλοτόφσκι, έχετε το λόγο. Δεν τον θέλετε όμως, σας ευχαριστώ. Κύριε Τέιλορ. Όχι, το συγγνώμη. Κύριε Τέλιτσκα. Κανένα πρόβλημα, κυρία Πρόεδρε, μην ανησυχείτε. Αν η κυρία Τέιλορ ήθελε πρώτη. Θα το θυμάμαι, αλλά δεν θα προσβληθώ. Τέλο πάντων. Θα είμαι σύντομο. Εκτιμώ το έργο του συγγετή μας, του κυρίου Σαλίνη. Έχει, ε, συνεργάστηκε πολύ καλά με τους Σκιώδης. Θεωρούμε ότι οι τροπολογίε που είχε υποβάλει η Άλντε έχουν ενσωματωθεί πλήρω. και εκτός αυτού γενικότερα ο εισηγητής έκανε μια ουσιαστική προσπάθεια να τροποποιήσουν το κείμενο της πρόταση της Επιτροπής με φιλοσοφία παρό, πολύ παρόμοια με την δική μας. Επομένως μπορούμε να υποστηρίξουμε την εκθέση αυτή. Σα ευχαριστώ. Και εμεί ευχαριστούμε κύριε Τελίτσκα. Κύριε Τέιλορ, έχετε το λόγο. Μάλλον από το, κούρεμα ήταν που μας μπέρδεψε η πρόεδρος, λέει ο κύριος Τέιλορ. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ κύριε Σαλίνη για την προετοιμασία του φακέλου. Οι πράσινοι καλωσορίζουν την κατεύθυνση που παίρνει. Συμφωνούμε επίσης και με τις συμβιβαστικέ τροπολογίες. Χαιρόμαστε επίσης που αναφέρεται η σημασία του να ε, ε, έχουμε τα μέγιστα κοινωνικο-οικονομικά ωφέλη από αυτά τα προγράμματα, το έγνος, το Γαλιλαίο, ιδιαίτερα όσον αφορά την, το περιβάλλον, η προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιήσουμε τα στοιχεία της παρατήρησης της γης από το Κοπέρνικος και αυτά να τα αξιοποιήσουμε για λόγους εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνολικά λοιπόν μιλώντα, υποστηρίζουμε το κείμενο του εισηγητή και τι συμβιβαστικές τροπολογίε και θα φανεί αυτό και στην ψήφο μα αύριο. Σα ευχαριστούμε κύριε Τέιλορ. Κυρία Αρ... Αρνατού. Σας ευχαριστώ. Κύριε εισηγητή, έχετε δίκιο. Το διάστημα που παραμένει στρατηγικής σημασίας θέμα και για την τεχνολογία. Παλαιότερα είχαμε τον ψυχρό πόλεμο μεταξύ της, των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης και είχαμε βρεθεί στο περιθώριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθώντας κάπως να ε, εισέλθουμε κι εμείς με πρωτοβουλία πρώτη της Γαλλίας και υπόδειγμα αυτής της ε, διακυβερνητικής ε, συνεργασίας, την οποία παρεπιπτόντως υποστηρίζει διαρκώς η ομάδα μας, ήταν το, η εκτόξευση των πυράβλων Αριάδνη 1 και 2 Σήμερα έχουμε και άλλους παίκτε. Έχουμε την Κίνα, σύντομα θα έχουμε την Ινδία στο διάστημα. Επομένω θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο να δίνει κίνητρα και να έχει επίσης και την αντίστοιχη χρηματοδότηση έτσι ώστε να δημιουργήσουμε και θέσεις εργασία, αλλά και να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στο, στην κούρσα του διαστήματο. Πιστεύουμε ότι διαφορετικά θα μείνει πίσω η Ευρώπη. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή πολιτική για το διάστημα γίνεται όλο και πιο περίπλοκη με όλο και περισσότερους ε, διαφορετικούς φορείς. Αντί αυτά τα θέματα να τα πραγματεύονται οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστεύουμε ότι είναι καλύτερα να παραμείνει στα χέρια των κρατών μελών, σεβόμενοι την κυριαρχία τους, αλλά επίσης και το δεδομένου ότι εκείνοι γνωρίζουν ε, και έχουν την εμπειρία σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης συζητήθηκε ένα ζήτημα με τη ε, διαχείριση των δορυφόρων και των συστημάτων Αριάδνη. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα σύστημα αριθμιστικό το οποίο να ε, ενθαρρύνει εκείνους που θέλουν ε, να δραστηριοποιηθούν στον τομέα του διαστήματος, τους ιδιώτες. Δεν έχουμε ένα σύστημα αντίστοιχο με το buy των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αγλάν Σαγλμό, πρόεδρος του, ε, του ομίλου Αριάδνη, πρόσφατα διακήρυξε, είπε ότι μόνο το 2 το 3, και με 3% της παγκόσμια αντίστοιχης αγοράς καλύπτεται από ευρωπαϊκές εταιρείε. Έχουμε έναν, μια προστατευτική πολιτική από τις Ηνωμένε Πολιτείε και κάτι το οποίο είναι, έχει δυσμενείς επιπτώσεις για την αεροναυπηγική βιομηχανία και διαστημική βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Γανονταλόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω το έργο που έκανε ο εισηγητής, ε, το οποίο είναι εξαιρετικό και δείχνει ότι χρειάζεται να έχουμε προτιμησιακή προτίμηση προς τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε έναν τομέα τόσο στρατηγικής σημασίας όπως το διάστημα. Σε αυτόν τον τομέα είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και οι άλλες μεγάλες δυνάμεις, να προτιμά και να, βοηθά τη βιομηχανία της. Θα ήθελα γι' αυτό και εμείς και άλλοι ε, συνάδελφοι έχουμε υποβάλει την τροπολογία για το άρθρο 25 προσπαθώντας να προστατεύσουμε ότι ε, στους στρατηγικούς ε, τομείς θα δίνονται προτιμήσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Κάτι αντίστοιχο έχουμε και με το άρθρο 114 με το, οποίο, 114, με το οποίο ζητούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει ένα πολυετές στρατηγικό σχέδιο για το διαστημικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτές είναι οι δικές μας τροπολογίες και ρωτώ από τους συναδέλφους αν είναι διατεθειμένοι να τις υποστηρίξουν. Σας ευχαριστούμε κύριο Δουκέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την εξαιρετική του εργασία. Η, η, η Κριστίνε προείπε αυτά που ήθελα να πω και εγώ μου κόβει τα φτερά δηλαδή. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να αξιοποιήσει τις ε, τεχνικές ε, του διαστήματος έτσι ώστε να εφαρμοστούν και επίγεια. Πέρσι είχαμε 150 δις ευρώ προστέμενη αξία για αυτές τις ε, δραστηριότητες. Είναι κρίμα λοιπόν να ε, αναπτύσσουμε διαστημικές δραστηριότητες και παράλληλα να μην μπορούν να καρποθούν και οι επίγειες δραστηριότητες. Βλέπουμε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις ε, κατέχουν ηγετική θέση με βάση εγχειρήματα ευρωπαϊκά. Επίσης, μας απείλησε ο θεσμικός χαρακτήρας, πρόσβαση στο διάστημα, αλλά τώρα ο εμπορικός χαρακτήρας ε, είναι αυτός που μας απειλεί. Είναι ένας άλλος τρόπος θεώρησης των πραγμάτων. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι εμπορικές επιχειρήσεις της Βόρειας Αμερικής έχουν κρατικές επιδοτήσεις και γι' αυτό ίσως θα πρέπει να μας απασχολήσει και στο δικό μας ε, σύστημα. Η κυρία Αρνοτού μας μίλησε ότι θα μπορούσαν τα κράτη-μέλη να ανταποκριθούν μόνο τους. Όμως ε, ως προς τους εκτοξευτές ε, στο διάστημα, εάν δεν υπάρχει Ευρώπη ως σύνολο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ευχαριστούμε κύριε Ρικέ. Η Επιτροπή τώρα, η Γενική Διεύθυνση, η Αρμόδια Γενική Διεύθυνση. Κύριε Σίλβα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Επιτροπή χαίρεται για τη συζήτηση που γίνεται εδώ στην Επιτροπή από όλες τις παρεμβάσεις που άκουσα. Θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι η έκθεση σαλίνη συμβαδίζει με τις προτάσεις μας. Η Επιτροπή θα ήθελε να βελτιώσει την πρόταση της, λαμβάνοντας υπόψη αυτά που άκουσα. Θα ήθελα να διευκρινίσω ορισμένα στοιχεία της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μην υπάρχουν λανθασμένες ερμηνείες. Εφαρμόζουμε το άρθρο 5 για να συμφωνήσουμε για, τις θεσμικές, για τα θεσμικά προαπαιτούμενα για τις εκτοξεύσεις στο διάστημα. Αυτό δεν αφορά εθνική κυριαρχία, Άρα τα κράτη-μέλη μπορούν να επιτρέψουν στην Επιτροπή να το κάνει. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι σήμερα για το πρόγραμμα ε, Γαλιλαίος δεν μπορούμε να εκτοξεύσουμε δορυφόρους παρά από ευρωπαϊκό έδαφος. Σε σχέση με τις άλλες ε, εκτοξεύσεις τύπου Κοπέρνικους γίνονται μέσω ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα μίας γαλλικής με βάση τις συμβάσεις που υπογράφονται έτσι ώστε να έχουμε μία ανταγωνιστική βιομηχανία εκτοξεύσεων. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό υπάρχει μία καινοτομία προτείνουμε 16 δις αλλά με μεγαλύτερη ευελιξία για να λάβουμε υπόψη τις ε, τεχνολογικές αλλαγές και σε επίπεδο εκτοξεύσεων έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε σε αυτές τις αλλαγές και να μπορέσει να καινοτομήσει και η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Μην ξεχνάμε ότι στο Horizon Europe θα υπάρξει ένα σημαντικό ποσό και εδώ θέλουμε την υποστήριξή σας έτσι ώστε να καινοτομήσουμε. Επίτα, αυτό που θέλουμε είναι να αυξήσουμε τις υπηρεσίες, δηλαδή να φτάσουμε στον Ευρωπαίο πολίτη με υπηρεσίες έτσι ώστε να ε, δεχτεί αυτό το διαστημικό οικοδόμημα και εμείς να είμαστε εταίρος σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι ένα ευρωπαϊκό σχέδιο γιατί κανένα κράτος μέλος από μόνο του δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει εάν θέλουμε να συγκρίνουμε με τις άλλες μεγάλες ε, δυνάμεις στο διάστημα κατακλείδη η συζήτηση που γίνεται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Οι συζητήσεις προχωρούν πολύ καλά. Τα δύο θεσμικά όργανα θα συμφωνήσουν και θα θέλαμε να βελτιώσουμε το πλαίσιο για να υπηρετήσουμε τον Ευρωπαίο πολίτη και εντός και εκτός Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε. Ο εισηγητής και πάλι ο κύριος Σαλίνη. Έχετε το λόγο. Υπάρχουν ε, διαφορετικά αιτήματα και προθέσεις. Αλλά εδώ θα πρέπει να δώσουμε ορισμένες απαντήσεις είτε στην γνωμοδότηση στις μεταφορές είτε στην εργασία μας στην Ήτρε επί του θέματος. Θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για ένα θέμα στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και από βιομηχανικής πλευράς ότι σε σχέση με τους εκτοξευτές, το άρθρο 5, εργαστήκαμε για να δημιουργήσουμε τους όρους και τις συνθήκες έτσι ώστε να είμαστε πρωταγωνιστές ως Ευρωπαϊκή Ένωση στην οικοδόμηση αυτής της στρατηγικής. Δεν θα πρέπει να υποπέσουμε σε μία προστατευτική αντίληψη το στρατηγικό σημείο ύψης της σημασίας εξαρτάται από το τελικό αποτέλεσμα που θα πρέπει να είναι μία στρατηγική σωστά οριοθετημένη, μία στρατηγική έτσι ώστε να κατέχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο ε, όχι μόνο κάταντι αλλά και άναντι και αυτό αφορά και τα συστήματα πλοήγησης όπως το Γαλιλαίο, όπου έχουμε μία διάρθρωση που είναι ανταγωνιστική, αλλά έχουμε και το θέμα χρήσης αυτών των υποδομών που θα πρέπει να δοκιμαστεί. Γι' αυτό Υπάρχει μεγάλη πίεση από τους οργανισμούς και επειδή έχουμε πολλές τροπολογίες, οι συμβιβασμοί κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτοί είναι οι κανόνες της αγοράς. Σε σχέση με τον προϋπολογισμό, το προείπαμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συνεργάζονται. Και τώρα στο ερώτημα για την τροπολογία 214 έχω αμφιβολίες γιατί νομίζω ότι τα ευρωπαϊκά προνόμια ε, είναι επαρκώς οριοθετημένα. Ευχαριστούμε κύριε Σαλίνη. Να σας υπενθυμίσω ότι η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το πρωί στις 9 η ώρα. Και μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης γνωμοδότηση ιδίας πρωτοβουλίας σχέση με τη στρατιωτική κινητικότητα. Ο κύριος Τίλτσκα είναι ο συντάκτης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Το θέμα αυτό δεν είναι καινούριο. Δεν το εξετάζουμε μόνο με αυτή τη γνωμοδότηση, αλλά είχε προκύψει και όταν εξετάζαμε τον κανονισμό Connecting Europe, του συνδέοντα στην Ευρώπη. Έχουμε 57 τροπολογίες, έχουν υποβληθεί. Και η ψηφοφορία θα γίνει επί τη βάση 6 συμβεβαστικών τροπολογιών. Θέλω θέλω να ευχαριστήσω τους συναδελφούς που υπέβαλαν τροπολογίες και έθεσαν κέρια ζητήματα. Γνωρίζω ότι η συζήτηση αυτή έχει δημιουργήσει κάποιες ανησυχίε σε ορισμένες πολιτικές ομάδες. Αυτό δεν περιορίζεται μόνο σε ορισμένα μέλη, αλλά σε μεγάλο μέρος της ομάδας. Και θα προσπαθήσω με τη γνωμοδότηση και τις συμβαστικές αυτήν να ανταποκριθώ σε αυτές τις ανησυχίες. Σημαντικά θέματα. Θα πρέπει να διευκρινιστούν οι διαδικασίες, οι κανόνες για τις διαδικασίες με τις οποίες θα χρησιμοποιούνται αυτά τα χρήματα για τη στρατιωτική κινητικότητα. Τι ακριβώς ορίζουμε ως στρατιωτική κινητικότητα. Και κάτι με το οποίο συμφωνώ με τον συνάδελφο Μαρινέσκου και το συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν το ζήτημα που είχε προκύψει και στο πλαίσιο του ΣΕΦ το να φροντίσουμε στρατιωτική κινητικότητα ή διπλής χρήση κινητικότητα να μην περιορίσει τους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την, ε, την, κινητικότητα μη στρατιωτική των πολιτών. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε βέβαια τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκριθεί όχι μόνο στο ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής αντιπαράθεσης, αλλά φυσικά και σε φυσικές καταστροφές, σε έκτακτες καταστάσεις ή άλλου είδους προβλήματα πολιτικής φύσεως στο εσωτερικό της. Νομίζω ότι αυτό τώρα φαίνεται ξεκάθαρα πια. Θα θέλαμε επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει τις προϋποθέσεις που τίθενται για να υποβληθούν προγράμματα στο TEN-T με στρατιωτικό χαρακτήρα. Ζητούμε ως δεσμευτική προϋπόθεση για να μπορεί ένα πρόγραμμα να χρηματοδοτηθεί από το ten να είναι διπλής χρήσεως και τονίζουμε επίσης ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα διασυνοριακά προγράμματα, στα προγράμματα τα οποία καλύπτουν τους, ε, ε, μετακινήσεις μεταξύ δύο κρατών μελών και είναι κάτι στο οποίο συμφωνεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύει ότι εκεί υπάρχουν και μεγαλύτερες ευκαιρίες. Χωρίς να πω περισσότερο σε λεπτομέρειες, συνολικά θα έλεγα ότι με τις συμβιβαστικές τροπολογίες έχουμε καλύψει τι τροπολογίε που υπέβαλαν οι συνάδελφοι. Βέβαια θα πρέπει να επιθυμίσω ότι δεν είμαστε επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή, είναι η ΣΕΝΤΕ. Εμείς κάνουμε μια γνωμοδότηση προς αυτήν και ε, επιδιώκουμε με την ψηφοφορία μας, με τη, τη δικιά μας γνωμοδότηση να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Επιτροπή Άμυνα και ασφάλεια. στα ζητήματα που είναι ε, ουσιαστική σημασία για την Επιτροπή Μεταφορών. Αυτά από πλευρά μου. Σα ευχαριστώ. Και εμεί ευχαριστούμε κύριε Τενιτσκά. Ήσασταν σαφέστατο. Κύριε Φαντεκάμπ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κατά πρώτον, Να πω ότι εκπροσωπώ την κυρία Μαριέσκου. Θα μιλήσω εκ μέρους της. Και να ευχαριστήσω τον κύριο Τελίτσκα και τους ασκιώδεις συζητητές για, την, για το εξαιρετικό τους έργο σε αυτή τη γνωμοδότηση που καθιστά σαφές ε, τους σκοπούς της Επιτροπής μας σε αυτόν τον τομέα ώστε να διαθέσουμε τα κονδύλια στους αντιδρόμους TNT για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου και να ότι θα έχουμε κατά τα σημαντικά ζητήματα. Δεύτερο, ότι στις κεντρικές του ΣΕΦΑ δεν έχουμε περίεργες διαδικασίες όπου εξαφανίζονται ε, κονδύλια ε, με συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το θέμα καλύφθηκε επαρκώς ε, στις συμβατιστικές προτάσεις. Έχει και το πρόγραμμα των εξοδότηση πράξεων, ο κύριος Τελίσκα, έχει το χρονοδιάγραμμα. Για να γνωρίζουμε τι κάνουμε από όλες τις πλευρές, κάτι που πρέπει να προσέξουμε και που περιέχεται στην τροπολογία 6 είναι η έμφαση στις νέες τεχνολογίες. Είμαι ένας απλός πολίτης Δεν σκέφτομαι τα τάγκς, αλλά την κυβερνασφάλεια, το ίντερνετ, τέτοια πράγματα. Το RTMS, το Σέζαρ. Ε, σε αυτό το θέμα θα πρέπει να σκεφτούμε νέους συνδυασμούς τεχνολογίας, ασφάλειας και μεταφορών. Γι' αυτό υποστηρίζω πλήρως ε, τις συμβαστικές σας ευχαριστούμε κυρία Γραπίνη, Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ισορροπημένη έκθεση. Συνεργαστήκαμε πολύ καλά και θετικά. Προσπαθούμε να έχουμε μία αποδοτική προσέγγιση αυτής της δαπάνης με διπλό στόχο και για την στρατιωτική και την πολιτική άμυνα και φτάσαμε σε ευρεία συνένεση. Ελπίζω να ψηφίσουμε αύριο τις τροπολογίες συμβιβασμού. Ε, θα ήθελα να συζητήσω ορισμένα άλλα στοιχεία με τον εισηγητή γιατί ας πούμε η τροπολογία 57 η δική μου προέβλεπε ότι τα κράτη-μέλη θα συνεργαστούν για την διασυνοριακή αποδοτικότητα. Δεν ξέρω γιατί απορρίφθηκε, γιατί εγώ πιστεύω σε αυτή τη συνδεσιμότητα μεταξύ κρατών μελών, ιδιαίτερα σε όμορες περιοχές. Δεν καταλαβαίνω γιατί απορρίφθηκε. Και βέβαια παραμένει το δίλημα της διπλής χρήσης υποδομών που πρέπει να αποκλεί τα λιμάνια και τα αεροδρόμια. Γιατί στα αεροδρόμια έχουμε και ειδικέ συνθήκες Γι' αυτό θα πρέπει να διαχωρίσουμε τη στρατιωτική υπόδομη από την πολιτική. Ε, ως προς τη στρατιωτική υποδομή την, ε, την χρησιμοποιούμε σε περίπτωση εμπόλεμης κατάστασης ή φυσικών καταστροφών. Δηλαδή και υπάρχει και πολιτική χρήση αυτής της υποδομής. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ζλωτόσκι έχει το λόγο. E, Συμφωνώ με τον κύριο Ταλίτσκα. Σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση, να σας ευχαριστήσω πολύ για την ε, καλή συνεργασία και υποστηρίζουμε το εγγραφό σας πλήρως. Ξεκάθαρο, πολύ εύγλωτο. Κύριε Τέιλορ, έχετε το λόγο. Thank you very Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι σύντομος. Ένας από τους ήταν ο Ντελόντε που δεν είναι εδώ, αλλά ήθελα να πω εκ μέρους του ότι δεν υποστηρίζουν την κατανομή των κονδυλίων υπό το CF γιατί το πρόγραμμα CF πρέπει να κινητοποιήσει έξυπνες, βιο, έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη, διευκολύνοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των αγαθών και των υπηρεσιών με την κατανομή της ιδιωτικής κινητικότητας, με την ε, συμπερίληψη σε αυτό το ε, ε, φάκελο, τότε ουσιαστικά θέτουμε σε κίνδυνο την μη στρατιωτική χρήση γιατί δεν υπάρχει εγγύηση ότι τα κονδύλια που θα πρέπει να πιστωθούν σε μη στρατιωτική χρήση, ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για στρατιωτική χρήση. Γιατί αυτά που αφορούν τη στρατιωτική χρήση έχουν να κάνουν με την οδοποιία και αν λάβουμε υπόψη ε, τις δεσμεύσεις που έχουμε για την ε, κλιματική αλλαγή θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την ανάγκη ότι πρέπει να ε, τηρήσουμε τις δεσμεύσεις αυτά ώστε να μπορέσουμε να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς. Άρα, ο φάκελος και η σωδική κινητικότητα αποτελεί πρόβλημα για αυτή την ε, επένδυση. Χρειάζεται να υπάρξει ε, ανάπτυξη των υποδομών που έχουν να κάνουν με μη στρατηγική χρήση για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες Και στην γνωμοδότηση αυτή θα θέλαμε να δούμε μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση όπου θα υπάρξει έμφαση και στην μη στρατιωτική χρήση. Ευχαριστούμε κύριε Αχνοτού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Τέλισκα για την έκθεσή σας. Οι τροπολογίε που έχουν υποβληθεί βεβαίω βελτιώνουν το κείμενο, όμω στην πραγματικότητα, κατά την άποψή μου, δεν απαντούν στο ουσιαστικό ερώτημα που ετέθηκε με μία από τι δικέ μα τροπολογίε, που είναι το εξή. Είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποκαταστήσει, υποκαταστήσει το ΝΑΤΟ. Έχουμε αυτό το στόχο η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή να μετατρέψει τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσει τις οδικές της ε, αρτηρίες για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ και να είναι σε θέση να το εξυπηρετήσει σε μια εντελώ υποθετική περίπτωση στρατιωτική σύρρηξης. Αυτό είναι κατά την άποψή μας στην ουσία το ζήτημα της ε, ερωτήματος που μας θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έρχεται το ζήτημα των φυσικών καταστροφών. Πολύ σπάνια όμω χρειάζεται η συμβολή του στρατού, αυτή είναι συμπληρωματική και σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε δει ουσιαστικά κάποιο πρόβλημα με, τις με, τα, τους δρόμους. Ε, ιδιαίτερα λοιπόν για τους εκείνους που δηλώνουν ειρηνιστές, αλλά και για εμάς, πιστεύουμε ότι το ζήτημα είναι βαθύτατο πολιτικό, ό,τι και να ψηφίσει κανείς και σας ζητώ να καταψηφίσετε την έκθεση. Η πρόεδρο, σας ευχαριστούμε και εμείς. Θα απευθυνθώ τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Κόλσον είναι ο πρόσωπός της. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα. Θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσει τον εισηγητή και το σύνολο της Επιτροπής σα για το έργο σας στο θέμα αυτό. Όσον αφορά τώρα τι τροπολογίες. Μετά μάλιστα και από την τελευταία τοποθέτηση του εισηγητή σας ε, που μας μίλησε για τις συμβιβαστικές τροπολογίες, μπορώ να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με την κατεύθυνση που παίρνουν. Ιδιαίτερα υποστηρίζουμε τη θέση που παίρνετε ότι σε καμία περίπτωση τα χρήματα αυτά δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις οι οποίες δεν έχουν και χρήση πολιτική. Οι επενδύσεις ε, οι οποίες θα ε, χρησιμοποιηθούν για τους διαδρόμους Και επίσης ότι αυτές οι, μετα... Ε, αυτές επενδύσεις θα πρέπει να βοηθούν τις πολυτροπικές μεταφορές, με όλους, όλες τις μεθόδους μεταφορές. Ράς. Θεωρούμε ότι αυτή η χρηματοδότηση μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, των εκτάκτων καταστάσεων, γενικά της πολιτικής προστασίας. Συμφωνούμε μαζί σας ότι η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει να ενισχύσει την πολυτροπικότητα και ιδιαίτερα τα διασυνοριακά έργα υποδομής. Επίσης συμφωνούμε μαζί σας ότι οι συγκεκριμένε ρυθμίσει, οι συγκεκριμένε προποθέσει θα καθοριστούν με πράξη κατεξουσιοδότηση πριν το 2019. Σε ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο τη Γενική Διεύθυνση ΜΟΥΒ για την παρέμβασή του. Κύριε Τελίτσκα, Τελίτσκα, έχετε το λόγο για να κλείσετε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω από το τέλος. Κάνατε λόγο από την πλευρά της Επιτροπής και κατανοώ τη θέση της ότι υπάρχει διαφορετική θεώρηση ανάλογα με την πολιτική ομάδα. Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που θα μπορούσαν κάποιοι να τα δουν ως κομμάτι πειρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει τις δικές της αρμοδιότητες και ικανότητες ναι, καταλαβαίνω την νίξη που κάνετε για την πολιτική προσέγγιση και θα χρησιμοποιήσω δικά μου λόγια ότι δεν το κάνουμε αυτό για να εξυπηρετήσουμε τον ΝΑΤΟ. Αντιθέτως, κάνουμε λόγο αποκλειστικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διαδικασίες είναι ξεκάθαρες και στα κείμενα που έχουν ήδη εγκριθεί. Θα έχουμε λοιπόν ένα ίδιο πλαίσιο ώστε να μην υπάρχουν εκτροχιασμοί. Επίσης κατανοώ ότι οι πράσινοι, κύριε Τέιλορ, έχουν τη δική τους τοποθέτηση. Είναι κρίμα ότι ο σκιώδης συγκητής δεν προσπάθησε να το συζητήσει αυτό το θέμα μαζί μου ώστε να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε και τη δική του άποψη. παρόλο που ήταν εύκολη η διαδικασία και υπήρξε συνένεση. Θα μπορούσαμε όμω ε, σε διμερέ επίπεδο να έχουμε μια διαβούλευση. Αυτό που δεν καταλαβαίνω, κύριε Τέιλορ, είναι γιατί κάποιοι από τους συναδέλφους μου από τους πρασίνους συνεχίζουν να έχουν την άποψη ότι, ότι παίρνουμε ε, κονδύλια από τον τομέα των μεταφορών. Το αντίθετο συμβαίνει και θα ήθελα να διαβάσουν ε, ό,τι υπάρχει διαθέσιμο οι συνάδελφοι, να δουν και το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οπότε, αν ε, ψηφίσετε ενάντια, θα είναι ενάντια στο να βάλουμε τον φάκελο των 6,5 εκατομμυρίων για τη στρατηγική χρήση στο CF. Στο CF. Άρα θα πείτε, ουσιαστικά θα πείτε στο κοινό ότι 6,5 δισεκατομμύρια δεν χρησιμοποιούνται και ότι θα χρησιμοποιηθούν στις μεταφορές αλλά ότι θέλετε να τα διοχετεύσουμε αλλού. Δηλαδή θα έχει αντίστροφο αποτέλεσμα η ψήφα σας αύριο. Αυτό όμως που σέβομαι είναι ότι οι πράσινοι έχουν μια τοποθέτηση. Κυρία Γραπίνη, που εκτιμώ τη συνεργασία της, είχαμε απευθεία επικοινωνία για να σας ε, δείξω ότι είναι σωστή αυτή η προσέγγιση στην τροπολογία 57 όπου κάνετε λόγους για συνεργασία των ε, κρατών μελών στις οδικές μεταφορές και στην ε, ελάφρυνση του διοικητικού κόστους σε διασυνοριακό επίπεδο. Είναι δύσκολη η γνωμοδότηση ώστε να καλύψει τα πάντα σε ένα περιορισμένο χώρο, όμως θεωρώ ότι αυτό θεωρείται δεδομένο και κατά δεύτερον κάνουμε ε, λόγω διασυνοριακή οδική μεταφορά και ένας λόγος που δεν θα είστε υπέρ είναι επειδή κάνουμε για οδικές μεταφορές. Πώς το γνωρίζετε αυτό? Θα δω την τροπολογία σας. Αυτός είναι ένας ο λόγος που υπάρχει εστίαση στις οδικές μεταφορές. Δεν αφορά μόνο στις οδικές μεταφορές, κύριε Τέιλορ. Αν ήθελα όμω βαρύ εξοπλισμό, δεν θα τον μετέφερα μέσω δια... με δική μεταφορά, αλλά με άλλους τρόπους. Επειδή έχω κάνει μου στο στρατό, θυμάμαι πολλά σχετικά με αυτό το θέμα για τα αεροδρόμια. Ναι, δεν θέλουμε να μπερδέψουμε τα στρατικά αεροδρόμια με τα μη στρατικά αεροδρόμια σε συγκεκριμένες περιοχές δεν υπάρχουν στρατητικά αεροδρόμιο. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες προσαρμογές ώστε να μπορεί ε, να μεταφερθεί ο βαρύς εξοπλισμός. Μπορεί να μην συμφωνείτε με την άποψή μας σε αυτό το θέμα. Θα έχουμε περισσότερες ευκαιρίες να το συζητήσουμε, να τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά και ανυπομονώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Τελτσκά. Κύριε Τέιλορ, ζήτησατε το λόγο. Ναι, για να δώσω κάποιε διευκρινήσει, κυρία Πρόεδρε. Καταλαβαίνω και χαίρομαι μάλιστα για τι παρεμβάσει του εισηγητή που λέει ότι δεν μπορεί να ξέρει, δεν μπορώ να ξέρω, δεν μπορώ να γνωρίζω. Γιατί όμω εγώ βασίζομαι στο που, ε, τι είδου έργα χρηματοδοτεί το Connecting Europe σήμερα. Δεν είμαι σκιώδης επί του θέματος αυτού, αλλά ευχαρίστως να ε, έχουμε την συζήτηση αυτή σε μία από τις ε, συναντήσεις των σκιωδών. Κύριο κύριος Ε, άρα λοιπόν ο κύριος Τέιλορ απλώς μεταδίδει που μεταφέρει πληροφορίες χωρίς να έχει γνώση. Αυτόν επομένως δεν θα σχολιάσω. Ευχαριστώ κύριε Τέλιτσκα. Υπενθυμίζω η ψηφοφορία αυτής της χρωμοδότησης της ίδιας πρωτοβουλίας θα γίνει αύριο. στι 9. Συνεχίζουμε με το τελευταίο μας ε, θέμα στην ημερησία διαταξή για σήμερα. Είναι το πρωτόκολλο που τροποποιεί την Ευρωμεσογειακή Συμφωνία Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και του Βασιλείου τη Ιορδανία αφετέρου, έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριο κύριος Keith είναι ο εισηγητή μας. Έχετε το λόγο. Για να μα παρουσιάσετε το σχέδιο σύστασή σα. Σας ευχαριστώ και πάλι, κυρία Πρόεδρε. Ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό το πρωτόκολλο, που θα συναυθεί μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωσης και του Χασιμητικού Βασιλείου της Ιορδανίας. Η πρότασή μου προ την Επιτροπή Μεταφορών είναι να δώσει τη σύμφωνη γνώμη τη για τη σύναψη του πρωτοκόλλου αυτού. Σα ευχαριστώ. Πρόεδρος, ήσασταν ε, ε, κύριε Κουτ. Θα είμαι σύντομος. Συμφωνώ και προτείνω να δώσουμε την έγκριση μας στο πρωτόκολλο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προταθούν τροπολογίες. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Je continue. Monsieur Telinska. Ευχαριστούμε κύριε Τέλισκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ συνεχίζω να μην έχω καταλάβει τι θα γίνει. Ε, μάλλον παρά το γεγονό ότι οι πράσινοι θα, θα λάβουν τη θέση που θα λάβουν στο πακέτο για την γενετικότητα, για αυτό το θέμα θα σας υποστηρίξω. Να ορίστε, λέει η πρόεδρος, που τα βρήκατε. Ζητάει κάποιος άλλος συνάδελφος το λόγο. Εάν όχι, ευχαριστώ πολύ. Θα σας υπενθυμίσω. θεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι. Να σας υπενθυμίσω ότι εδώ πρόκειται για διαδικασία σύμφωνης γνώμης επομένως τροπολογίες μόνο επ' αυτού είναι δεκτές. Επί του θα δώσουμε δηλαδή συμφωνή γνώμη ή όχι. Εάν δεν υπάρχει κάποιο άλλο συνάδελφο, θα συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μα και κλεισμένων των θυρών, στη συνεδρίαση συντονιστών. Και τα υπόλοιπα μέλη, με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών θα τα πούμε αύριο το πρωί, 9 η ώρα, για τις ψηφοφορίες. Τώρα θα περάσουμε στη συνεδρίαση των συντονιστών. Και θα κάνουμε και μια μικρή διακοπή για να σταματήσει το web streaming και για να φύγουν όσοι δεν δικαιούνται να βρίσκονται στην αίθουσα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.